πόρους. Ελπίζω λοιπόν ότι χάρη σε αυτών των προδιαγραφών θα μπορέσουμε κάποια μέρα να συζητήσουμε για το τέλος αυτής της κατάστασης στην Καμπανία. Ο κύριος Κονσολίνο δεν είναι εδώ, αλλά ε, υπάρχει άλλος ομιλητής σχετικά με την καμπάνια. Όχι, τότε έληξε και το θέμα αυτό τα πρακτικά θα υποβληθούν στη, για αποδοχή στην επόμενη συνεδρίαση. Ε, τα ψηφίσματα που έχουν υιοθετηθεί θα αναφερθούν και έλξη συνεδρίαση.